Οι αρμόδιες αρχές της ελληνικής δημοκρατίας μου απέστειλαν έτοιμα για την άρση της βουλευτικής αλυσίας του Γιώργου Κίρτσου για τις ε, ποινικές διαδικασίες του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου των Αθηνών εναντίον του. Η εξέταση του θέματος θα γίνει από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και από τις αρμόδιες αρχές του